αύριο. Πάμε τώρα στο επόμενο σημείο της τη διατάξεως που είναι η κοινή συζήτηση για την απαλλαγή της χρήσης 2013. Ο κύριος Τσαρνέτσκι είναι ο συντάκτης της δεύτερης έκθεσης. Η δεύτερη δε και η τρίτη έκθεση ακριβώ έχουν συνταχθεί από τον κύριο Τσαρνέσκη, στον οποίο και θα δώσουμε το λόγο. Μπορείτε να μας παρουσιάσετε τις εκθέσεις. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, πρόκειται για πάρα πολύ σημαντική συζήτηση. Κρίμα που η συζήτηση αφήγεται τόσο αργά. Μέσα στη νύχτα γιατί συνήθως τέτοια ώρα είναι ώρα για να βλέπει κανείς θρίλερ και αστυνομικά, αλλά τέλος πάντων εδώ μιλούμε για χρήμα. Για χρήμα πρέπει να περάσει από έλεγχο, από εποπτεία, ούτω ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα να προστατεύσουν τα συμφέροντα των φορολογουμένων. Μιλούμε τώρα για το Ινστιτούτο της Βουδαπέστης που ασχολείται με την καινοτομία και την τεχνολογία. Έχουμε τώρα αυτόν τον οικονομικό έλεγχο όσον αφορά κάποιες ε, υποτροφίες. Θέλουμε επίσης να βελτιωθεί το σύστημα χορηγήσεως κάποιων πιστοποιητικών και θέλουμε να τροποποιηθούν οι διαδικασίες και οι προβλεπόμενες διατάξεις. Θα πρέπει να δούμε όμω αυτή η πιστοποίηση, πώ θα ρυθμιστεί στι λεπτομεριές τη, πώς θα γίνονται επίση οι διαγωνισμοί, υποβολή προσφορών κλπ. Επομένω, ε, θα πρέπει να σας πω με μία φράση ότι πρόοδο έχει επιτευχθεί. Τώρα, όσον αφορά την ε, νομιμότητα των ε, συναλλαγών, των σχετικών με τις υποτροφίες αυτές, τα πράγματα έχουν πάει καλά το Δέλεγκτικό Συνεδρίο για δεύτερη συνεχή χρονιά υπέβαλε την αιτιολογημένη έκθεση. Θα πρέπει να μην ξεχάσουμε ότι περίπου 87% των ε, δαπανών ήταν αντικείμενο πιστοποίησεων των ε, οικονομικών ελεγκτών. Πρόκειται επομένως για μια διαδικασία που θεωρείται ότι έχει κινδύνους παρατυπιών. Επομένως, θα πρέπει να σας πω ότι αυτές οι δύο ε, αιτιολογημένες γνώμες οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι στο παρελθόν τα πράγματα δεν λειτουργήσαν όπως θα έπρεπε. Επομένως, να ελέγξουμε το τι έχει γίνει και να διαπιστώσουμε κατά πόσον το Ινστιτούτο έχει εφαρμόσει τους κείμενες διατάξεις. Τώρα, όσον αφορά το Artemis και το ENIAC. Δεν μπορούμε να μπούμε τώρα ε, στις λεπτομέρειες γιατί ήδη έχουν γίνει σχετικοί έλεγχοι και τώρα όσον αφορά το Συμβούλιο είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει επανειλημμένα και στις ε, εκθέσεις που συνέταξα νωρίτερα το Συμβούλιο. Είναι ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο. Επομένω, έχει ευθύνη, ευθύνη δημοκρατική λειτουργία έναντι των πολιτών. Θα πρέπει ό,τι κάνει να αναλογεί στα όσα προβλέπονται από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Όμως, έχουμε κάποια θέματα διότι το Συμβούλιο πάρα πολύ συχνά δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματά μας για παροχή εξηγήσεων. Και επομένως δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει το ότι ε, λέμε όχι στην ε, απαλλαγή προς το Συμβούλιο. Επομένω, θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι καθόλου όμορφο. Παιχνίδι μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Θα πρέπει αυτό το παιχνίδι να λάβει τέλος. Όμως χρειάζεται να υπάρχει πολιτική βούληση από πλευρά του Συμβουλίου. Κύριε Στυλιανίδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σιγητά. Εκπροσωπώ εδώ την αγαπητή αντιπρόεδρο, την κυρία Γεωργίευα η Κομισιόν σημειώνει τις ε, προτάσεις της Επιτροπής ε, Δημοσιονομικού Ελέγχου προς την Ολομέλεια για να δοθεί απαλλαγή στην ε, κοινή επιχείρηση Άρτεμις και την κοινή επιχείρηση για τα ηλεκτρονικά την έννοια και για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας και να αρνηθεί την απαλλαγή στο Συμβούλιο για το Οικονομικό Έτος 2013. Ε, η Κομισιόν με χαρά σημειώνει πως η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου συμφωνεί πως το κοινό εγχείρημα που θα διαδεχτεί τις επιχειρήσεις Άρτεμις και ENIAC έχει προβεί σε ενέργειες για να ανταποκριθεί στις παρατηρήσεις της αρχής προπολογισμού και άρα σκοπεύετε να δώσετε απαλλαγή για το έτος 2013. Το ΕΝΙΑΚ και η Άρτεμις επέδειξαν πως η ΣΔΙΤ χρησιμοποιώντας ένα τριμερές μοντέλο με χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης Κρατών Μελών και της ε, βιομηχανίας μας δίνει την δυνατότητα να φτιάξουμε τσίπ ε, κορυφαίας τεχνολογίας και με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας μεταξύ άλλων. Έτσι, η βιομηχανία στην Ευρώπη έχει ένα σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αποκτά δυνατότητα να αναπτυχθεί όπως κατέδειξε η υψηλή επένδυση που υπήρχε στην σύμπραξη αυτή. Και οι δύο πρωτοβουλίες είχαν μεγάλο βαθμό μόχλευσης. Κάθε δημόσιο ευρώ κατέληξε σε επένδυση τουλάχιστον τριών ευρώ από τον κλάδο στις δύο πρωτοβουλίες. Το ενιακ και η Artemis άρα είναι μια μοναδική ευκαιρία και ένας αποτελεσματικός τρόπος για την βιομηχανία, τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστούν στενά και έτσι δημιουργείται μια κρίσιμη μάζα για ηλεκτρονικά συστήματα και μέρη που έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης. Οι πρωτοβουλίες χρηματοδοτούν κάθε χρόνο πάνω από 3.000 κορυφαίους Ευρωπαϊ... Ευρωπαίους μηχανικούς και ερευνητές. Και η δουλειά τους βοηθάει να ε, διατηρηθούν τουλάχιστον 80.000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη κάθε χρόνο στο πρόγραμμα πλαίσιο για τον ορίζοντα 2020 το ENIAC και η Artemis οι δύο κοινέ επιχειρήσεις πάνε σε μια νέα κοινή επιχείρηση για ηλεκτρονικά μέρη Excel όπως λέγεται όπου βρίσκουμε μια δομική λύση για ελέγχους εκ των υστέρων και επαλήθευση των νέων δαπανών στο σχέδιο ψηφίσματος ε, ζητάτε από την Κομισιόν να κάνει μια αξιολόγηση για να ε, δει εάν οι δραστηριότητε ε, της Αρτέμιδας και του ΕΝΙΑΚ μπορούν να τύχουν απαλλαγής εμείς λοιπόν σκοπεύουμε να το κάνουμε αυτό με τον κανονισμό Excel που προβλέπει πως η Κομισιόν θα κάνει μια ενδιάμεση αξιολόγηση του Excel που θα περιλάβει την τελική αξιολόγηση του ΕΝΙΑΚ και της Αρτέμιδος μέχρι την 30 Ιουνίου 2017. Θα κάνει επίσης μια ξεχωριστή αξιολόγηση ε, τώρα για τα ίδια έργα ξανά σημαίνει πως θα έχουμε υπερβολικό διοικητικό βάρος ε, και για τους ε, δικαιούχους και για την Κομισιόν. Τέλος να πω πως η Κομισιόν θα στηρίξει και θα δώσει σύμβουλες στο εγχείρημα Excel για να ανταποκριθεί σε αυτά τα οποία θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας έχει κάνει σημαντικές βελτιώσεις στους τομείς που ανέφερε η απόφαση του Κοινοβουλίου του Απριλίου για την νομιμότητα και την κανονικότητα των συναλλαγών. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο έχει βελτιώσει την μεθοδολογία του ελέγχου. Υπάρχουν επίσης νέες κατευθυντήριες γραμμές για την προκήρυξη και τις προμήθειες και άρα το ποσοστό σφάλματος ε, είναι μόλις 0,9%. Επίσης, ε, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας έχει λάβει μέτρα για να βελτιώσει τον προγραμματισμό και την εποπτεία. Τέλος, σημειώνουμε πώς ο κύριος Γκοβίντα που κέρδισε φέτος, ε, ο κύριος Γκοβίντα Αμπετουάη που κέρδισε φέτος το βραβείο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κοινοτομίας και Τεχνολογίας επελέγει ακριβώς ε, για να βραβευτεί και στο πλαίσιο των 30 ε, πολλά υποσχόμενων επιστημόνων κάτω των 30 ετών και γι' αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς σκοπό έχει και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κοινοτομίας και Τεχνολογίας η Κομισιόν λυπάται για το ότι ε, δεν ε, μπορέσαμε να βρούμε μια λύση για την απαλλαγή του Συμβουλίου για τις δύο δημοσιονομικές αρχές που πλέον διαφωνούν εδώ και έξι χρόνια. Η Κομισιόν θεωρεί πως τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να συνεργαστούν για να λειτουργήσει ομαλότερα η διαδικασία. Ελπίζουμε λοιπόν να επιληθεί το ζήτημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ευχαριστώ, Μαρινέσκου, για ένα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτά τα κοινά εγχειρήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά όσον αφορά την έρευνα αλλά και την ανάπτυξη. Διότι εδώ υπάρχουν πάρα πολύ ψηλά ποσά σαν πρικοδότης και θα πρέπει επομένως και η διαχείριση να είναι αντίστοιχη. Οπότε πρέπει να δούμε ότι αυτές οι κοινέ επιχειρήσεις ε, διέπονται από κάποιες ε, καθυστερήσεις, αυτό είναι τις προηγούμενες χρήσεις και οπότε και ήρθαμε ή στην βελτίωση φέτος γιατί θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με την αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Ελληνικού Συνεδρίου για το 2014. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ψήφισε υπέρ, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν έρθουμε στο θέμα του 2014, γιατί χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια και πιο προσεκτική ανάλυση. Θα πρέπει επομένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα πει για το ΕΝΙΑΚ ε, περισσότερε λεπτομέρειε και τέλο πάντων. Ε, έχει υποσχεθεί ότι θα το πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογία επίση έχει κάνει ήδη μια διαδρομή. Θα πρέπει να καταλάβουμε πώ λειτουργεί και να έχουμε την προκαταρκτική έκθεση, γιατί αυτό είναι θέμα του χρήματο των ε, φορολογουμένων. Τώρα, όσον αφορά την απαλλαγή προ το Συμβούλιο, θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα συγκεκριμένα. Και ε, ξέρω ότι είχαμε αρνητική στάση πολύ καιρό γιατί έχουμε ευθύνη εναντί των πολιτών. Θα μπορούσε να πει κανεί ότι η διαδικασία τη ε, απαλλαγή είναι ένα ανέκδοτο. Ένα λεπτό Βόν. Okay. Uh, uh, thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω για την απαλλαγή του EIT. η σκιώδης εισηγητής για τον οργανισμό αυτό. Να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για την ε, συνεργασία του. Ξέρετε, αρνηθήκαμε να δώσουμε απαλλαγή για το EIT για διάφορους λόγους. Καταρχάς για το ε, στατιστικό, το δείγμα σφάλματος 3%. Μετά βρήκαμε λάθη στις διαδικασίες για τις προμήθειες και διάφορα άλλα λάθη που έχουν να κάνουν με τα νούμερα που έχουν να κάνουν με το προσωπικό. Έκτοτε έχει σημειωθεί πρόοδος από το EIT. Μας την έχουν αναφέρει αυτή. Και επίσης την έχω, έχω επισκεφτεί αυτόν τον οργανισμό. Είδα την πρόοδο από μόνος μου και μπορώ να το βεβαιώσω. Το error rate έχει πέσει από το 3% στο 2,9%. Έχουν νέες διαδικασίες για την προμήθεια και νέες διαδικασίες για την αξιολόγηση του προσωπικού. Και αυτό ε, θα βοηθήσει στη μείωση του προσωπικού. Επομένως είμαι υπέρ της απαλλαγής του EIT να δοθεί και όταν έχουμε και την έκθεση από το Ελεκτικό Συνέδριο για το 2014 τότε θα δούμε πραγματικά την ουσιαστική πρόοδο που έχουν ε, καταβάλει. Ε, Αλή για δύο λεπτά. Παρακαλώ. Thank you, Mr. Chair, Mr. Commissioner, Mr. Chernetsky, colleagues. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τον Απρίλιο αναβάλαμε την απόφαση απαλλαγή του Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομία Τεχνολογία για την Οικονομική Χρήση 2013. Στα τέλη του Ιουνίου λάβαμε μια έκθεση από το EIT ε και μας έδινε η έκθεση αυτή πληροφορίες. Και με βάση αυτή τη νέα έκθεση αντλούμε τα εξή συμπεράσματα. Ως προς την νομιμότητα και την νομοφροσύνη των συναλλαγών, το Ινστιτούτο έχει βελτιώσει την ποιότητα των πιστοποιητικών ελέγχου. Η χρήση νέας μεθοδολογίας έχει βελτιώσει την ποιότητα εκ των προτέρων και εκ των υστέρων επαληθεύσεων όλα ήδη πληρούν τις αντίστοιχους κανόνες για τις προμήθειες και το Ινστιτούτο πλέον έχει δυνατότητες εσωτερικού ε, οικονομικού ελέγχου. Ως προς τον προϋπολογισμό και τα οικονομικά υπάρχουν θετικές αλλαγές, γίνεται καλύτερο σχεδιασμός, καλύτερη εποπτεία, παρακολούθηση και έχει βελτιωθεί η δυνατότητα ε, απορρόφησης των δικαιούχων. Και ως εκ τούτου Πέραν από τις διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε θετικές εξελίξεις και ως προς το σχέδιο δράσης του Ινστιτούτου. Στα τέλη του 2015 περιμένουμε να ολοκληρωθούν αυτές οι δράσεις. Άλλωστε, επίκειται ειδικό, δημοσίευση ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου που θα ε, μας δώσει τη δυνατότητα να καταλάβουμε κατά πόσο πραγματικά το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο αυτό έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει την καινοτομία και την τεχνολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να τα συζητήσουμε με τις σχετικές πανεπιστημιακές κοινότητε. Είναι θετικέ οι αλλαγέ και θέλουμε να απαλλαγεί ο διευθυντή είμαστε υπέρ αυτή τη πρόταση για την οικονομική χρήση 2013. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόλτες για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ. Εγώ θα επικεντρωθώ στο ζήτημα της απαλλαγής του Συμβουλίου. Έχουν περάσει έξι μήνες από όταν αναβάλαμε την απαλλαγή του Συμβουλίου. Και σήμερα πάλι συζητάμε το εάν ε, θα μας δώσει στοιχεία για τα οικονομικά του το Συμβούλιο. Η διαδικασία της απαλλαγής είναι υποχρεωτική για όλα τα θεσμικά όργανα και το Συμβούλιο δεν αποτελεί εξαίρεση. Πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν το πώ υλοποιείται ο προπολογισμό του όπω ακριβώ και των υπολείπων θεσμικών οργάνων. Πώ είναι δυνατόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην ε, μπορεί να δει τον προπολογισμό του Συμβουλίου εδώ και τόσα χρόνια. Και τόσα χρόνια να μην βλέπουμε καν ε, τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου εδώ πέρα όταν συζητάμε το ζήτημα. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν πως θα υπάρχει λογοδοσία και θα πρέπει επιτέλους να υπάρχει και κάποια αξιοπιστία του Συμβουλίου. Είμαι λοιπόν πεπισμένος πως ε, δεν αρκεί, δεν ακούν πλέον οι παρενέσεις προς το Συμβούλιο. Οπότε οι πράσινοι έφεραν μια τροπολογία που για πρώτη φορά ε, έχει μια δημοσιονομική επιφύλαξη για το Συμβούλιο έτσι ώστε να μην μπορούμε να δώσουμε απαλλαγή και να τιμωρήσουμε την ε, συμπεριφορά αυτή και για τον προπολογισμό του 2016. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το θάρρος του που λέει ότι πρέπει να δώσουμε απαλλαγή ε, για τον προπολογισμό του 2013 για το Συμβούλιο. Ε, σπάνια βεβαίως ασκείται κριτική εδώ μέσα σε άλλο θεσμικό όργανο. Υπάρχει πράγματι πρόβλημα επικοινωνίας. Δεν απαντά στις ερωτήσεις το Συμβούλιο. Ερωτήσεις για δαπάνες, για δεσμεύσεις, για τα κτίρια, το Residence Palace, για την διοικητική οργάνωση, οπότε θα ήθελα να πω πως ε, εγώ επενώ το θάρρος το ασυνήθιστο του εισηγητή, αλλά δεν είναι τόσο ασυνήθιστο, γιατί η απαλλαγή δεν δόθηκε ούτε το 2009, 10, 11, 12, 2013 και για το 2013 μιλάμε και ακόμα δεν έχουμε απαντήσεις. Δηλαδή Είτε πιστεύει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα, είτε όχι. Εάν λοιπόν κανείς θα πιστεύει, είναι ντροπή να αγνοούν έτσι το Κοινοβούλιο. Αν δεν πιστεύει κανείς όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς τα πράγματα είναι τα γνωστά και συνήθη. Σας ευχαριστώ. Σντετσόφσκι για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Ήδη από την αρχή της θητείας μας είπαμε ξεκάθαρα ότι δεν θα ανεχθούμε λάθη, ε, σφάλματα, ε, ποσοστό και συντελεστές σφαλμάτων και λαθών στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, το ιστορικό του Ινστιτούτου ήταν πολύ κακό και στην εφαρμογή του προϋπολογισμού και στην αμοιμότητα των επιχορηγήσεων που λάμβανε δεν, ήταν, δεν είχαν την ικανότητα να κάνουν προληπτικούς ελέγχους, εξάντε. Και γενικά όλη η διαχείριση ήταν πολύ, πολύ αδύναμη και γι' αυτό αποφασίσαμε να αναστείλουμε τις ελεκτικές δραστηριότητες. Ωστόσο, όταν ανέλαβε η νέα διοίκηση, το Ινστιτούτο έκανε τεράστιες προσπάθειες και γι' αυτό αποφασίσαμε υπέρ της απαλλαγής και θα συνεχίσουμε να τους παρακολουθούμε και να τους εποπτεύουμε. Έχουν βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, στηρίζω την απαλλαγή και στο βαθμό που θα συνεχίσει το Ινστιτούτο να αντιμετωπίζει τα προβλήματά του και να προσπαθεί να τα λύσει, όλα θα είναι καλά. Αυτό όμως έρχεται σε ευρία αντίθεση με το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο έχει αποτύχει και δεν τους δίνουμε απαλλαγή. Και νομίζω ότι τώρα είναι η μπάλα στην πλευρά του γηπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ε, μας βοηθήσει να λύσουμε το πρόβλημα. Ο κύριος Μπαλτσίτης, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Νομίζω ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο όσον αφορά το πρόγραμμα δράσης και την εφαρμογή του. Και έτσι νομίζω ότι θα μπορέσουμε ε, αυτά τα οποία έχει ζητήσει το ελληνικό συνέδριο να τα διορθώσουμε όσον αφορά δηλαδή, τον οικονομικό έλεγχο. Όσον αφορά επίση την πιστοποίηση ποιότητος, έχουμε επίση και ανταλλαγή πληροφοριών και ανταλλαγή των ε, αρίστων πρακτικών. Έχουμε χάραξει μια πολιτική και την έχουμε βελτιώσει όσον αφορά την ε, σύγκρουση συμφερόντων και όλα αυτά αφορούν και το Άρτεμις και το ΕΝΙΑΚ. Πρόκειται για μια κοινή επιχείρηση και θα πρέπει όλα αυτά τα νέα στοιχεία να εφαρμοστούν και οπότε πρέπει να δώσουμε την απαλλαγή. ενάμιση από το κύριο Ντόιτς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μία απαλλαγή για το Συμβούλιο δεν είναι τίποτα το καινούριο. Εδώ και χρόνια αγνοεί τις ερωτήσεις μας το Συμβούλιο. Είναι η πέμπτη φορά που αρνούμαστε να δώσουμε απαλλαγή. Δεν είναι ποτέ παρόντες όταν συζητάμε την απαλλαγή του. Δεν απαντάνε στις ερωτήσεις μας. Δεν μας δίνει τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την διαδικασία της απαλλαγής. Δεν έχουμε πληροφορίες ε, για το τι γίνεται με την πολιτική των κτηρίων, πόσα είναι τα έξοδα, τα αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να δούμε την οικονομική διαχείριση, άρα δεν μπορούμε να λάβουμε κάποια σοβαρή απόφαση. Το Συμβούλιο δεν σέβεται την ε, διαδικασία η οποία ισχύει για όλα τα θεσμικά όργανα. Οπότε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υποστηρίζει την πρόταση του εισήγητη. Σας ευχαριστώ, Σάρβαμα, που, που είναι, δεν είναι στην η κυρία Γκρέσλε λοιπόν για ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η απαλλαγή είναι κάτι το οποίο προβλέπεται στη συνθήκη. Και ακριβώς αυτή την ώρα περιμένουμε για να εξετάσουμε και εμείς ε, πώς ξοδεύονται τα λεφτά. Κύριε Επίτροπε, θετικά αυτά τα οποία είπατε για τις κοινέ επιχειρήσεις, αλλά θα πρέπει λίγο η Κομισιόν να το πάρει πάνω στο θέμα. Χρειάζεται κάποια εποπτεία και πάντα απορούμε με τα προβλήματα σε αυτούς τους μικροσκοπικούς προϋπολογισμούς. Είναι μικροσκοπικοί και θα πρέπει να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια από ό,τι βλέπουμε. Να έρθω τώρα στο Συμβούλιο. Είναι σκάνδαλο το ότι το Συμβούλιο δεν ε, ε, καταδέχεται να ε, μας επιτρέψει να ελέγξουμε το τι κάνουμε τον προπολογισμό του ενώ ελέγχει όλα τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να σχηματίσουμε μια συνολική εικόνα και θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή το Συμβούλιο να αφαιρέσει αυτό το αγκάθι από τη σχέση μας. Είναι πια γελία η κατάσταση. Ευχαριστώ. Μπόγκοβιτς για ένα λεπτό. Μικρό. I Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Είναι μια φυσιολογική διαδικασία η απαλλαγή και σε εταιρείε ιδιωτικού δικαίου αλλά και όσον αφορά ε, δημόσιους φορείς. Στη μία περίπτωση είναι η μέτοχη και στην άλλη είναι η τα στελέχη της, ε, ε, της, ε, του, του δημόσιου οργανισμού. Οπότε έχουμε προκειμένου αυτές, αυτούς τους οργανισμούς, το ΕΙΤΑΤΑΦ, ΕΕ, το Άρτεμις, έχουν γίνει διάφορες βελτιώσεις τελευταία, οπότε και τηρήθηκαν οι οδηγίες. Ποιο είναι τώρα το πρόβλημα. Το Συμβούλιο ακόμη είναι απρόθυμο να αναλάβει τις ευθύνες πενάντι του Κοινοβουλίου. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο λέει ο συγκητή και να μην παράσχουμε την απαλλαγή στο Συμβούλιο. Α ελπίσουμε στο μέλλον το Συμβούλιο να βελτιώσει την ε, συμπεριφορά του. Και τώρα για το Catch the Eye, λέει ο Πρόεδρο. Έχει ο κύριο Μαριά το λόγο. Τον έχετε. Κύριε Πρόεδρε, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η δημοκρατική λογοδοσία προ του φορολογουμένου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο με βάση τα άρθρα τρία δεκαέξι τρία και τρία δεκαεννιά συνθήκης λειτουργίας ευρωπαϊκής ένωσης έχει το δικαίωμα χορήγησης απαλλαγής για κάθε τομέα του προϋπολογισμού της ένωσης χωριστά άρα και για το τμήμα ευρωπαϊκό συμβούλιο συμβούλιο. όμως το συμβούλιο θεωρεί ότι είναι κράτος εν κράτη ότι είναι περάνω κάθε ελέγχου γι' αυτό και επί σειρά ετών εξακολουθεί να μην απαντά στις ερωτήσεις του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου οι δαπάνες του συμβουλίου πρέπει να ελέγχονται όπως ελέγχονται οι δαπάνες των υπολείπων οργάνων της ευρωπαϊκής ένωσης και όμως το συμβούλιο επιδεικνύει έλλειψη συνεργασίας αρνείται να δώσει αναλυτική γραπτή εξήγηση για το συνολικό ποσό πιστώσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά του κτηρίου residence palace. στηρίζω λοιπόν την έκθεση του κυρίου Τσαρνιέτσκι, που δεν χορηγεί απαλλαγή στο γενικό γραμματέα του συμβουλίου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ευρωπαϊκού συμβουλίου και συμβουλίου για το. 2013. ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σιγητά, όπως ξέρετε εκπροσωπώ εδώ την συνάδελφό μου, την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα και θα ήθελα άρα να σας ευχαριστήσω που δίνετε την ευκαιρία να πάρω τον λόγο για την κοινή συζήτηση για τις απαλλαγές του Συμβουλίου, τις κοινέ επιχειρήσεις και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας. Και βεβαίως ε, καλωσορίζουμε τις προτάσεις σας για να δοθεί απαλλαγή στις κοινές επιχειρήσεις και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας. Οι κοινέ επιχειρήσεις έχουν ε, κάνει σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου και η Κομισιόν θα συνεχίσει να τους δίνει συμβουλές και στήριξη στις προσπάθειες τους για να ανταποκριθούν σε αυτά τα οποία ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τσαρνέτσκι έχει τον λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριοι συνάδελφοι. Είναι κρίσιμη η στιγμή αυτή στη ζωή μου τώρα που σας μιλάω. Να σας πω στο τέλος γιατί το λέω αυτό. Πάντως, να απαντήσω σε όσα έχουν αναφερθεί. Είναι αλήθεια ότι ήδη έχουμε βγάλει κίτρινη κάρτα ε, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογία. και νομίζω ότι με το δίκαιο μας το κάναμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έκανε βήματα πρόοδου και άρχισε να λειτουργεί καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Τώρα, όσον αφορά το Συμβούλιο, τι έγινε. Πριν από έξι μήνες Κάναμε το ίδιο και με το Συμβούλιο. Δείξαμε την κίτρινη κάρτα, αλλά δεν υπήρξε κανένα είδου ε, απόκριση. Τίποτα. Καμία αντίδραση. Οπότε συμφώνησαν όλες οι πολιτικές ομάδες ότι πάνω από τις επιμέρους διαφορές μας αυτό είναι απαράδεκτο. Για πέμπτη χρονιά αντιμετωπίζουμε τέτοιο πρόβλημα με την Ρωσία και ο κύριος Όλτες καλά τα είπε ότι άλλα περιμένουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Πρόκειται περί σκανδάλου. Ξέρω ότι αυτή η έκφραση είναι πολύ έντονη, αλλά είναι ακριβής, διότι το Συμβούλιο αρνείται να συνεργαστεί. Και αυτό επανειλημμένα. Πολύ σωστά αναφέρθηκε ότι αυτή η ιστορία δεν έχει τέλος. Θα πρέπει μόνος και εμείς να σταθούμε συνεπής, είναι και θέμα τιμής για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να δείξουμε υπευθυνότητα έναντι των Ευρωπαίων, έναντι των ψηφοφόρων μας. Δεν είναι δυνατόν να υποχωρήσουμε, να ενδώσουμε, θα πρέπει να πιέσουμε το Συμβούλιο, να το αναγκάσουμε, να ανταποκριθεί. Θέλουμε να είμαστε εταίροι, να υπάρχει διάλογος. Ε, τώρα, γιατί σας είπα ότι πρόκειται για πάρα πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή μου, γιατί μόλις τώρα έμαθα ότι ο γιος μου εξελέγει βουλευτής για δεύτερη φορά στο Πολωνικό Κοινοβούλιο. Με μεγάλη μου χαρά, εγώ σας το ανακοινώνω. Συγχαρητήρια του λέει και ο πρόεδρος του κυρίου Τσαρνέτσκι. Τέλειωσε εκείνη η συζήτηση και πρόκειται να ψηφίσουμε για αυτές τις εκθέσεις αύριο. Θα μπορούσατε να επεκταθείτε με κάποια αφορμή επερώτηση, αλλά τέλος πάντων. Συγχαρητήρια και πάλι.